Έχουμε δύο εισηγητές, την κυρία Γκροστέτ και τον κύριο Τάνα Σέσκου. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη, την κυρία Γκροστέτ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω οι συνάδελφοι να πρόλαβαν να φτάσουν στην αίθουσα της Ολομελίας γιατί πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τους ασκιώδης συγητές και το επιτελείο του Επιτρόπου Ανδριουκάητης που συνεργάστηκε μαζί μου για το θέμα αυτό. Πάνω από χίλιε τροπολογίε, ε, πάνω από 150 άρθρα και παράγραφοι. Κολοσιαίο έργο Τιτάνιο που το, που το επιτελέσαμε από κοινού με πνεύμα συνεργασία και συμβιβαστική λύση και διαλλακτικότητα. Χαίρομαι ιδιαίτερω γι' αυτό. Άλλωστε ήταν απαραίτητο αυτό το πνεύμα ε, γιατί ήταν σημαντικά τα δικηβέματα αυτής της ε, νομοθετικής αναθεώρησης. Και ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός ε, Υγείας μας προειδοποιεί ότι κινδυνεύουμε να βυθιστούμε σε ένα κόσμο μετά, μετά των αντιβιωτικών, όπου η μικροβιακή αντοχή θα δημιουργήσει περισσότερους θανάτους από τον καρκίνο. Θα πρέπει λοιπόν να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του. Η καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής θα πρέπει να ξεκινήσει από την εκτροφή των ζώων από την κτηνοτροφία. Θέλουμε λοιπόν να απαγορεύσουμε την προληπτική χρήση των αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία. Να περιορίσουμε τις μαζικές θεραπευτικές αγωγές σε συγκεκριμένα ζώα και επίσης να ε, απαγορεύσουμε τη χρήση σημαντικών ε, αντιβιωτικών μόνο σε ανθρώπινη χρήση και να απαγορεύσουμε και την διαδικτυακή πώληση εμβολίων, αντιβιωτικών και ψυχότροπων ουσιών. Επίσης έτσι θέλουμε να περιορίσουμε ε, το, την ποσότητα των αντιβιωτικών που φτάνει στα πιάτα των καταναλωτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μειώσουμε το θεραπευτικό πλωστάσιο των κτηνιάτρων. Είναι υπεύθυνοι επαγγελματίε οι κτηνίατροι και του έχουμε εμπιστοσύνη. Και άλλωστε είναι και αρμόδιοι και πλέον κατάλληλοι για να επιλέξουν την καλύτερη θεραπευτική αγωγή ανάλογα με τι περιστάσει. Και ο κανονισμό αυτό το στόχο έχει, να διευκολύνει το έργο των κτηνιάτρων. Δεν θέλουμε να ρυθμίσουμε υπέρ των δέων το επάγγελμα αυτό που ήδη έχει δείξει την προσήλωσή του σε μεγαλύτερη αυστηρότητα και ηθική σοβαρότητα. Υπάρχει και το θέμα της διαθεσιμότητας ε, των ε, ε, φαρμάκων στην κτηνιατρική αγορά. Για να προσπίσουμε λοιπόν και να διαφυλάξουμε την υγεία των ζώων θα πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα των, θεραπευτικών αγωγών και να περιορίσουμε την θέση σε εμπορία ή την αδειοδότηση των φαρμάκων. Θα πρέπει επίσης να θαρρύνουμε την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Γι' αυτό και είναι πολύ φιλόδοξη η την αδειοδοτηση των φαρμακων θα πρεπει επισης να ενθαρρυνουμε την ερευνα και τεχνολογικη αναπτυξη στον τομεα αυτο γι αυτο και ειναι πολυ φιλοδοξη η εκθεση μου προτείνει το εξή. Προτείνει επέκταση ε, κάποιων περιόδων ε, εμπορική αποκλειστικότητα, ιδιαίτερα των φαρμάκων για τα ίσονο σημασία είδη, προκειμένου να δημιουργήσουμε σημαντικά κίνητρα για την έρευνα. Μερικές φορές ε, οι διοικητικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα επαχθείς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση και αυτό δημιουργεί τροχοπέδι στη θέση σε εμπορία καινοτόμων προϊόντων. Γι' αυτό και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδιατυπώσαμε κάποιες διατάξεις προκειμένου να θεσπίσουμε ένα νέο σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης που θα είναι πιο ελαστικό, πιο αποτελεσματικό και λιγότερο γραφειοκρατικό. Με ταχύτερες διαδικασίες θα έχουμε μια πιο έγκαιρη και άμεση αντίδραση των εργαστηρίων σε περίπτωση ζωνόσων επιζωτιών χωρίς να διακυβεύουμε ή να υπονομεύουμε τις προδιαγραφές μας ασφάλειας και ποιότητας που είναι από τις υψηλότερες του κόσμου. Τέλος, ο νέος αυτός κανονισμός θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξυπηρετήσει τους εκτροφείς, τους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς που αντιμετωπίζουν ήδη γνωστές δυσκολίες και είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι από το κείμενο του κανονισμού. Η νομοθετικές λοιπόν διατάξεις δεν θέλει να στιγματίσει τους γεωργούς και κτηνοτρόφους, αλλά να τους βοηθήσει να φροντίσουν καλύτερα τα κοπάδια τους. Επίσης, Συνεργάστηκα με την Επιτροπή Γεωργίας και με τα Συνδικάτα Εκτροφέων ώστε οι κανόνες αυτοί να εφαρμοστούν πολύ εύκολα επί τόπου και να μην προσθεθούν στο γραφειοκρατικό άκθος που ήδη τους βαρύνει. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να πω ότι είχαμε ένα τριπλό εδώ στόχο. Προστασία τη υγεία των ζώων και άρα και τη υγεία των ανθρώπων. Καταπολέμηση τη μικροβιακή αντοχή ε, και ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα ε, τη κτηνοτροφίας και της, ε, του κλάδου των κτηνιατρικών φαρμάκων. Φαίνονται ίσως αντιφατικοί εκ πρώτης όψης στόχη, στόχοι, αλλά καταφέραμε να τους ε, συνδυάσουμε και να τους συμφιλιώσουμε στην ομοθετική αυτή έκθεση. Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο, το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο, το μπαλάκι βρίσκεται στην πλευρά του Συμβουλίου και περιμένουμε ανυπομονησία τα σχόλια των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ κυρία Συγκήτρια. Το λόγο τώρα έχει ο δεύτερος ε, εισηγητής, ο κύριος Σταναζέσκου, τον οποίο όμως δεν βλέπω στην αίθουσα. Οπότε θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Ανδριουκάητης. Thank Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, χαίρομαι που μας προσφέρετε ευκαιρία να συζητήσουμε τις ε, προτάσεις αναθεώρησης ε, της νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να ε, διατίθενται περισσότερα τέτοια φάρμακα και να ενισχυθεί ουσιαστικά η ευρωπαϊκή δράση για να αντιμετωπιστεί η μικροβιολογική αντοχή. Ξέρω ότι το θέμα απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως πολύ καλά γνωρίζετε συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες σας. Ξέρω ότι η Επιτροπή ΕΝΒ στις 17 Φεβρουαρίου ενέκρινε αυτή την έκθεση με συντριπτική πλειοψηφία και δράτω με τις ευκαιρίες για να συγχαρώ την κυρία Γκροστέτ για την πάρα πολύ καλή δουλειά της, την κατέθεσε και έγκαιρα. Τη συγχαίρω επίσης για την αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Γκροστέτ κατόρθωσε να επιτύχει υποστήριξη σε 39 τροπολογικές που καλύπτουν την αναθεώρηση της πρότασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει κυρίως τις προσπάθειες που έγιναν για επικοδομητικές προτάσεις και εναλλακτικέ λύσεις αναφορούν ε, στη σήμανση, στην αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, φαρμακοεπαγρύπνηση και τέλος ε, ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τους στόχους ε, της πρότασης. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην αναθεώρηση του κανονισμού 726. Ε, Αυτή η αναθεώρηση είναι απολύτως απαραίτητη ε, για να υπάρχει αποκεντρωμένη χορήγηση αδειών. Είναι αυτός ο πρωταρχικός στόχος. Ο δεύτερος είναι να υπάρχει εναρμόνιση με τον ε, κανονισμό που προηγήθηκε και η Επιτροπή στις 17 Φεβρουαρίου ενέκρινε αυτές τις προτάσεις. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τανασέσκου για τη δουλειά του ως εισηγητής αυτού του θέματος που σφραγίστηκε με την έγκριση της ε, έκθεσης από συντριπτική πλειοψηφία. Η Κομισιόν έχει καταβάλει προσπάθειες να βελτιώσει την πρόταση και να λάβει υπόψη τη τη ιδιομορφή του κτηνιατρικού τομέα. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω ότι η συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, την Επιτροπή για τα δύο αυτά θέματα ήταν περισσότερο από αγαστή. Εμείς ε, θα προσπαθήσουμε να παραμείνει αυτό και στο μέλλον, τα θέματα να τελεσφορήσουν το συντομότερο δυνατόν και είμαι πεπισμένος ότι θα υπάρξει πρώτη ανάγνωση. Αυτό είναι ευκταίο και είμαι πεπισμένος ότι η ψηφοφορία θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για το Συμβούλιο για να επιταχύνει τις εργασίες του. Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι υπέρ του αγώνα κατά του MR. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει κάποιες πρακτικές λύσεις και νομίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ένα πρόγραμμα δράσης ε, για να ενισχυθεί αυτή η διαδικασία που αφορά στην μικροβιακή αντοχή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, να φέρουμε κοντά εμπειρογνώμονες ε, από όλους τους τομείς στον κτηνιατρικό τομέα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο μέσα στα σύνορά της όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η δική σας λοιπόν η δουλειά, η επικοδομητική αυτή δουλειά αποτελεί σημαντική συνεισφορά για να επιτύχουμε ε, στους στόχους μας. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για τις προτάσεις που κατέθεσε και ε, για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει ε, τη συμμετοχή του στην συνεχιζόμενο αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρξουν καινούργια μέτρα που να αφορούν στην μικροβιακή αντοχή και αυτά να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, προσοχή σας και προσβλέπω στο να ακούσω τις απόψεις των αξιότιμων μελών. Ευχαριστώ Επιτροπέ. Ο κ. Στανασέσκου ήρθε, οπότε ως δεύτερος συγητής λαμβάνει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν να ξεχωρίσουμε την αδειοδότηση για τα ε, κτηνιατρικά ε, φάρμακα από αυτήν για τα φάρμακα προς ανθρώπινη κατανάλωση, για την ανθρώπινη υγεία. Ο ισχύων κανονισμός έπρεπε να αλλάξει Μιλάω για τον 726 του 2004. Χρειαζόμουν περισσότερα στοιχεία και για λόγους ε, σαφήνειας, δεδομένου ότι όλα τα άρθρα αφορούσαν ε, όλα τα άρθρα που αφορούσαν τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν συμπεριληφθήκαν ε, στις καινούριες διατάξεις. λέμε ότι ο ΕΟΦ είναι ο υπεύθυνο για την ε, κεντρική αδειοδότηση των φαρμάκων και για τα φάρμακα για την ανθρώπινη υγεία και για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Η έκθεση εγγυάται το ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τους ε, δημοσιονομικούς κανονισμούς. Έχουμε λοιπόν πλέον όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τον προπολογισμό του ΕΦ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ε, στην Επιτροπή ΕΜΒΗ η έκθεση υπερψηφίστηκε μεγάλη πλειοψηφία οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προχωρήσει ε, για τον καθορισμό των τελών. Αναγνωρίζουμε το ρόλο του ΕΟΦ σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα. Χρειάζεται ο οργανισμός να συνεργαστεί με ιδρύματα ιατρικής τεχνολογίας προκειμένου να ε, ανταλλάξουν επιστημονικά δεδομένα. Η, ο ΕΟΦ θα πρέπει να δίνει στα κράτη-μέλη επίσης να παρέχει στην, ε, στα κράτη-μέλη ανάλυση για την ε, χρήση των φαρμάκων για, ανθρώπινη, για την ανθρώπινη υγεία τα οποία θα τα χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη εθελοντικά όταν θέλουν ε, στον, στις αποφάσεις τους για, τις, για τον καθορισμό των τιμών και των ε, επιστροφών ε, ε, της συμμετοχής του κράτους στην κοινωνική ασφάλιση. Ω ε, συνσηγητή, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γκροστέτ και του άλλου συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία μα. Νομίζω ότι με τις εκθέσεις μας βελτιώσαμε τις συνθήκες χρήσης των κτηνιατρικών προϊόντων. Ε, Επίσης βελτιώνουμε τις αγωγές που χωρίζονται στα ζώα και το πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας. Θέλουμε να αυξήσουμε την πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και να δώσουμε στους κτηνιάτρους περισσότερες εναλλακτικές λύσεις, περισσότερες επιλογές. Επιπλέον, ε, μιλάμε και για τις περιορισμένες αγορές. Η κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρμακών, κτηνιατρικών προϊόντων στα κράτη-μέλη θα πρέπει να βελτιωθεί μέσω καλύτερου συστήματος αδειοδότησης και καλύτερων ε, μεθόδων λιανικής τα Αυτά τα κτηνιατρικά φάρμακα μπορούν να πολλούνται ε, στο ίντερνετ με, με συγκεκριμένες βέβαια εξαιρέσεις για κάποιες κατηγορίες. Αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στον τομέα των φαρμάκων για την ανθρώπινη υγεία. Στηρίζουμε τα κρατημέλη ε, σε ό,τι αφορά τις, on, την online συνταγογράφηση. Ε, τα, θα πρέπει να ρυθμίσουμε το θέμα των αντιβιωτικών ε, και για την ανθρώπινη υγεία αλλά και για την ιατρική χρήση δεν, ε, θα πρέπει, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά για προφυλακτικούς λόγους ε, και προληπτικούς λόγους. Ε, θα πρέπει να βρούμε επίσης τρόπους για να καταπολεμήσουμε τη μικροβιακή αντοχή. Όλοι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών αρχών, των κτηνιάτρων και των αγροτών. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τώρα της Επιτροπής Γεωργίας, το λόγο έχει ο κύριος σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, την κυρία Γκροστέτ ε, και τον κύριο Τανασέσκου για το πολύ αξιόλογο έργο τους. Είχαμε 1111 τροπολογίες. Χάρη στη βοήθειά σας όμως καταλήξαμε σε εξαιρετικές συμβαστικές τροπολογίες που συνοψίζουν ε, τις πολυάριθμες αυτές τροπολογίες. Σημαντικός ο κανονισμός αυτός, όχι μόνο για την ευημερία των ζώων, για την υγεία των ζώων και για την ανάπτυξη των κτηνιατρικών φαρμάκων, αλλά και για την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι σημαντικό να περιορίσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών φαρμάκων. Και η ομαδική θεραπευτική αγωγή, η προφυλακτική χρήση αντιβιωτικών να μην επιτρέπονται. Χαίρομαι επίσης που έχουμε και ορισμό για το ποιος δικαιούται να συνταγογραφεί κτηνιατρικά φάρμακα, πώς θα χρησιμοποιούνται και πώς θα αντιμετωπιστεί και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Βρέθηκε πραγματικά η χρυσή τομή, η σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των καταναλωτών και της παροχής κινήτρων στο φάρμα, στον τομέα κτηνιατρικών φαρμάκων, προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα αλλά και να προωθήσουν τα γενώσιμα. Επίση, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη μικροβιακή αντοχή και να προστατεύσουμε ταυτόχρονα και το περιβάλλον μα. Έτσι θα έχουμε εύκολη πρόσβαση σε αποτελεσματικά φάρμακα που θα παράγονται και θα χρησιμοποιούνται με τρόπο που δεν θα απειλεί ούτε τη δημόσια υγεία, ούτε την υγεία των ζώων, ούτε των περιβάλλων. Γι' αυτό και η Άλντε υποστηρίζει ε, ολόθερμα τις δύο εκθέσεις και ελπίζω να μας μιμηθούν και άλλες πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Πόλτσακ και πάλι από την Επιτροπή Γεωργίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μόνο ένα λεπτό, γι' αυτό και θα περιοριστώ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τανασέσκου, γιατί έκανε δεκτέ πολλέ τροπολογίε τη Επιτροπή Γεωργία και τις συμπεριέλαβε στην έκθεσή του. Είχα κάποιες αφιβολίες σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως με την δομή της πρότασης και της προτάσεις για τον ΕΟΦ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, και για το θέμα των τελών και κατά πόσο θα πρέπει να καθοριστούν αυτά μέσω μιας εκτελεστικής πράξης. Η απόφαση για τον προσδιορισμό ε, του ύψου των τελών θα πρέπει να υπάρχει στη διαδικασία συναπόφαση με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μην αποτελεί το αντικείμενο μια απλή εκτελεστική πράξη. Στον κανονισμό αναφέρονται σε πολλά σημεία κτηνιατρικά φάρμακα και προϊόντα και γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί ο ρόλος και να αποσαφινιστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων καθώς και η προσπάθεια συγκέντρωσης των διαδικασιών σε ένα κεντρικό φορέα θα πρέπει, επαναλαμβάνω, τα τέλη να είναι προσιτά και σχετικά φθηνά. Αυτά και τώρα περάμε στη συζήτηση με προσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Τσίριο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, κυρίως ε, τη Νάλπο Γκροστέτ, με την οποία εργαστήκαμε αρκετά, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην Επιτροπή ε, καταθέσαμε τροπολογίες αλλά τελικά ε, καταλήξαμε και σε συμβιβασμούς. Ε, κατά την άποψή μου αυτό που πρέπει να εξάρουμε είναι ότι εδώ μιλάμε για νέους κανονισμούς και πολύ σύντομα ε, θα αρχίσει κανείς να φοβάται ότι η Ευρώπη θα επιβάλλει νέους κανόνες σε ένα τομέα που είναι ήδη πολύ επιβαρημένος με γραφειοκρατία. Μιλάμε για τους τομείς της γεωργίας και των κτηνοτρόφων. Αυτή είναι μια παραδοχή που δεν ισχύει όμως, ισχύει το αντίθετο. Εδώ πρόκειται για κανόνες οι οποίοι όμως δοκιμάστηκαν στην πράξη και δεν θα συνεπάγονται περαιτέρω ε, επιβάνηση της γραφειοκρατίας και είναι κυρίως ε, κανόνες που θα οδηγήσουν σε εναρμόνιση στην Ευρώπη. Ε, έτσι λοιπόν με αυτή την περίπτωση, με αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι όταν μιλάμε για τους κτηνοτρόφους μιλάμε κατά κύριο λόγο για το γάλα. Όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γονατίσει το γάλα, βιώνει μια πίθανη κρίση. Αυτοί λοιπόν οι κανόνες θα βοηθήσουν τον τομέα του γάλακτος γιατί είναι κανόνες οι οποίοι ε, θα ισχύουν για όλους ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα δηλαδή ε, όσοι παράγουν γάλα και εκτρέφουν ζώα θα έχουν να αντιμετωπίσουν τους ίδιους κανόνες γιατί αν οι κανόνες δεν είναι οι ίδιοι και δεν γίνονται σεβαστοί με τον ίδιο τρόπο τότε μπορεί κάποιος να πουλάει γάλα πιο φτηνά από την τιμή που ισχύει στην Ιταλία ας πούμε. Έχουμε λοιπόν ένα νέο κανονισμό, μπαίνουν όλοι κάτω από την ίδια ομπρέλα και αυτό θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημα. Ε, είναι άλλο ένα μήνυμα ότι δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, πρέπει να τις στηρίξουμε γιατί βιώνουν σκληρή και αδυσόπιτη κρίση. Πολύ ωραία. Η κυρία Κάντενμπαχ, ε, η επόμενη ομιλήτρια. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή την εβδομάδα ήδη γκρίναμε τον ε, νόμο περί της ε, προστασίας της υγείας ε, των ζώων. Αυτό άπτεται και της δημόσιας υγείας. Πρέπει να υπάρχει καλή πρακτική ε, να γίνεται σωστή χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων. Αυτή η προσεκτική χρήση των φαρμάκων νομίζω ότι επισημάνθηκε και από την κυρία Γκροστέτε και από άλλους εισηγητές. Είμαι λοιπόν ευγνώμων που τελικά κατέστη δυνατόν να ε, καταλήξουμε σε συμβιβασμούς διότι οι συμβιβασμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι είναι απαραίτητο η υγεία των ζώων και η υγεία των ανθρώπων να αντιμετωπίζεται κάτω από το ίδιο πρίσμα. Ε, Αυτά λοιπόν τα φάρμακα ε, θα πρέπει όμως να διαχωρίζονται άλλα τα φάρμακα για τους ανθρώπους και άλλα για τα ζώα. Βέβαια να προάγουμε την καινοτομία, να συμβάλλουμε έτσι ώστε κυρίως εκείνοι που χορηγούν αυτά τα φάρμακα να μην είναι εκείνοι που τα πουλάνε, να μην κερδίζουν από αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το θέμα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Επίσης να ρυθμίσουμε την πώληση ε, μέσω διαδικτύου, να απαγορεύσουμε την πώληση αντιβιωτικών από το διαδίκτυο. Αυτό το πακέτο θα βελτιώσει πάρα πολλά, θα υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, θα προάγεται η καινοτομία και όλα αυτά θα συμβάλλουν έτσι ώστε να ενισχυθεί ο αγώνας κατά της μικροβιακής ε, αντοχής. Κάτω από αυτό το πρίσμα είμαι πεπισμένη ότι ακολουθούμε το σωστό δρόμο και ελπίζω το ε, θέμα αυτό η έκθεση να υπερψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία. Ο κύριος Πιέχα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση της κυρίας Γκροστέτ και η έκθεση του κυρίου Τανασέσκου είναι αξιόλογες και τις δέχομαι με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Μάλιστα έγιναν σε ένα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας και αναζήτησης συμβαστικών τροπολογιών. Ε, είναι δύσκολο αυτό το θέμα και δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία, γιατί ζητούμενο δεν είναι μόνο η υγεία των ζώων και η προστασία της υγείας των ζώων αλλά ταυτόχρονα η προστασία της υγείας και των ανθρώπων, η ασφάλεια των τροφίμων αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Έχουμε διάφορες πτυχές της ασφάλειας. Έχουμε την ασφάλεια των ζώων, την ασφάλεια της, ε, του ανθρώπου που χρησιμοποιεί τα κτηνετρικά φάρμακα, την ασφάλεια του καταναλωτή των τροφίμων, την ασφάλεια του, ε, του ασθενούς ε, που θα πρέπει να το προστατεύσουμε από τη μικροβιολογική αντοχή. Για να μην μιλήσουμε και για την ασφάλεια του περιβάλλοντος, για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών και χαίρομαι που αυτό είναι ο στόχος του κανονισμού. Επίσης θα πρέπει να δούμε τη διαφορά μεταξύ προφυλακτικής και μεταφυλακτικής χρήσης ε, των ε, αντιβιωτικών και να γίνει σωστή διάκριση για να αποφευθεί η προφυλακτική χρήση και η χρήση ως αγωγή ελέγχου. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια διοδότησης, τα χαρακτηριστικά της διαφήμισης. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Η διαφήμιση και η διανομή τέτοιων προϊόντων μέσω του διαδικτύου δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το θέμα της προστασίας των δεδομένων γιατί κακές διατάξεις στον τομέα αυτό μπορούν να, να καταβαραθρώσουν οποιοδήποτε ερευνητικές προσπάθειες. Επίσης ε, καταθέσαμε πολλές τροπολογίες για την ε, έκθεση του κυρίου Τανασέσκου. Έχω αμφιβολίες για τα λεγόμενα ομοιοπαθητικά φάρμακα που περιορίζονται, ε, προέρχονται από ιδεολογικά περισσότερα κριτήρια παρά επιστημονικά πορίσματα. Ε, ακόμη και για τους ανθρώπους χρειάζεται πίστη για να είναι αποτελεσματικά τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Ε, για τη χρήση των ομοιοπαθητικών στην, στα ζώα έχω πολύ σοβαρές εμφωλίες για την αποτελεσματικότητά τους. Κύριε Πιέχα, έχετε μπλε κάρτα από τον κύριο Τζάνι. Τη δέχεστε? Βεβαίως. Κύριε Τζάνι, έχετε μισό λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία και κύριε Πιέχα που δέχεστε την μπλε κάρτα. Είπαμε και συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ αξιόλογες οι εκθέσεις. Έχω να σας κάνω μια ερώτηση. Ε, θεωρείτε ότι στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει στενότερη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και να παρακολουθεί καλύτερα την όλη διαδικασία. Μα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εμπίπτει περισσότερες αρμοδιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που, γιατί έχει εκτελεστικό χαρακτήρα. Θα πρέπει φυσικά να έχουμε βεβαιότητα για την ασφάλεια των κτηνιατρικών φαρμάκων και των, ε, φαρμάκων για την ανθρώπινη χρήση. Σε πολλές χώρες ο ίδιος οργανισμός επιλαμβάνεται και των κτηνιατρικών φαρμάκων και των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση. Γιατί υπάρχει αλληλεξάρτηση ε, και αλληλεπίδραση σε ό,τι αφορά τα φάρμακα αυτά. Γι' αυτό και συμφωνώ να είναι κεντρικό ο φορέα και για, τα, τις δύο κατηγορίε φαρμάκων. Ευχαριστώ. Κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Τανασέσκου και την κυρία Γκροστέτ. Με αυτές τις δύο εκθέσεις ε, θα βελτιωθεί κάτι πολύ σημαντικό που αφορά στην μικροβιακή αντοχή ε, για την οποία συζητούμε διαμακρών. Ε, στην έκθεση Τανασέσκου γίνεται λόγος ε, για τα φάρμακα, για τον άνθρωπο και για τα ζώα. Αυτά πρέπει να, είναι, να διαχωρίζονται. Να γίνει και σχετική προσαρμογή στη συνθήκη της Δισαβόνας Επίσης ε, και τα τέλη προς αυτό τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ λογικά. Αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι, κυρία Γκροστέτ, ότι πράγματι πρέπει να ασχολούμεθα προφύλαξη εκ των υστέρων θεραπεία ε, κυρίως όσον αφορά την προφύληξη, να μην υπάρχουν πλέον κρίσιμα αντιβιωτικά, ε, να μην δίδονται φάρμακα μέσα από τις ζωοτροφές, το πολύ πολύ αν πρόκειται το ζώο να εγχειριστεί. Επίσης τα αντιβιωτικά να χορηγούνται στα ζώα μόνο από κτηνιάτρους. Το βρίσκω σημαντικό και αυτό που είπε ότι ε, κάποια αντιβιωτικά ε, πρέπει να περιορίζονται μόνο στον άνθρωπο ή για τον άνθρωπο ε, για να είναι και αποτελεσματικά οποτεδήποτε χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, αν ένα αντιβιωτικό δεν υπάρχει σε ένα κράτος μέλος, μπορεί ένα άλλο κράτος μέλος να πάρει κάτι παρεμφερές. Και σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορούν να δοθούν στα ζώα ακόμα και ανθρώπινα αντιβιωτικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γενικές γραμμές ισχύει ότι θα πρέπει κάθε φορά να χορηγείται το αντιβιωτικό που πρέπει να χορηγηθεί. Εγώ σε αντίθεση με τον προλαλήσαντα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να επιτρέπεται και ομοιοπαθητική στα ζώα. Βεβαίως τώρα θέλετε, μπορούμε να διαφωνήσουμε αν αυτό έχει αποδειχθεί επιστημονικά ή όχι, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επιτρέπονται τα πάντα για να θεραπεύονται τα ζώα χωρίς να προκαλούμε την ενίσχυση της μικροβιακής αντοχής. Κυρία Κιλώνεν, 1,5 λεπτό. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές αλλά και όλους τους ε, συναδέλφους ε, για το πνεύμα συνεργασίας που έδειξαν. Όταν μιλάμε για κτηνιατρικά φάρμακα μιλούμε και για αντιβιωτικά και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο εν λόγω ο κανονισμός ασχολείται επίσης και με την ε, διαθεσιμότητα ε, των φαρμάκων και όχι μόνο με διοικητικά θέματα. Όταν πολλούνται και συνταγογραφούνται αντιβιωτικά θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Η αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν καταργούσε στην πράξη τη δυνατότητα ε, εθνικής μείωσης χρήσης αντιβιωτικών στα ζώα. Αυτό ε, θα μας δυσχέρνε στη Φιλανδία διότι θα χαλάρωνε το σύστημά μας. Χαίρομαι που κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Επιτροπή φροντίσαμε έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν τη δυνατότητα να έχουν αυστηρότερους κανόνες. Τα αντιβιωτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον μάλλον στη Φιλανδία τα αντιβιωτικά πολλούνται μόνο με συνταγή. Γι' αυτό το λόγο και το κρέας και το γάλα στη Φιλανδία δεν είναι γεμάτα αντιβιωτικά. Όταν τα... Ε, ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Να ευχαριστήσω τους πάντες και τους συνεισηγητές. Ευχαριστώ. Χάουσλινγκ, 1,5 λεπτό. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια και τους συναδέλφους. Δουλέψαμε εξαιρετικά μαζί. Προφανώς και βελτιώσαμε την πρόταση της Επιτροπής. Νομίζω πρέπει να επισημάνουμε ότι πρέπει ε, κάτι να κάνουμε γιατί υπάρχει μια κατάσταση απαράδεκτη δηλαδή ε, στην ε, κτηνοτροφία κυρίως κατά την πάχυνση χορηγούνται πάρα πολλά αντιβιωτικά απαράδεκτο αυτό υπάρχει το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής και στην Ευρώπη έχουμε 26.000 θανάτους από τη μικροβιακή αντοχή ε, σας λέω αυτό οφείλεται και στην εκτροφή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ασχοληθούμε με την προφύλαξη, τη μεταφύλαξη, ε, να μην χρησιμοποιούνται ε, τόσα πολλά αντιβιωτικά στα ζώα γιατί ε, το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται και η συγκεκριμένη έκθεση επιλαμβάνεται του προβλήματος για να χρησιμοποιούνται λιγότερα αντιβιωτικά. Και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Να συζητήσουμε και για εφεδρικά αντιβιωτικά, ε, τα οποία ε, όμως αφορούν τον άνθρωπο και εδώ δεν πρέπει να κάνουμε συμβασμούς. Επίσης, να βελτιωθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη συλλογή των δεδομένων. Δεν είναι ικανοποιητική η τράπεζα δεδομένων, πρέπει να εξοικειωθούμε και με ε, των αντιβιωτικών ε, επίσης και με την παραγωγή τους. Ένα θέμα θέλω να επισημάνω. Ο συνάδελφος από το ECR δυστυχώς έχει φύγει. Κοιτάξτε τι, τα ομοιοπαθητικά δεν πρέπει να τα περιφρονούμε, να τα αναγνωρίσουμε και ό,τι είναι εναλλακτική λύση των αντιβιωτικών να τα προβάλλουμε. Γι' αυτό εγώ ε, συμφωνώ με τη σχετική τροπολογία έτσι ώστε ε, να μην απαγορεύεται η ομοιοπαθητική στα ζώα. Ευχαριστώ. Ο κ. Πεντιτσίνη, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το κείμενο αυτό της Επιτροπής ΕΜΠΗ είναι ένα πολύ καλό κείμενο και ευχαριστώ τη Σνάλφο Γκρουστέτ που επέτρεψε σε όλες τις ομάδες να καταθέσουν τροπολογίες έτσι ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω το κείμενο της Επιτροπής. Θέλω να πω ότι η Κομισιόν ε, υπογράμμισε επανειλημμένα το βασικό στόχο αυτής της έκθεσης που είναι να ε, προκαλέσει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, να βελτιωθεί η λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Εμείς πιστεύουμε ότι το θέμα το νομοθετικό σε σχέση με τα φάρμακα πρέπει να έχει κύριο στόχο να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και την ευζοία των ζώων. Ήδη υπάρχει κάποια έκθεση πρωτοβουλίας για την ασφάλεια των ασθενών. Εκεί επισημάναμε την μικροβιακή αντοχή και στα κτηνιατρικά φάρμακα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί ε, η πολυτέλεια των αντιβιωτικών ε, περιορίζεται μόνο σε ζώα ε, που είναι άρρωστα. Κατά την άποψή μας πρέπει να βρούμε νέα αποτελεσματικά αντιβιωτικά και μπορούμε να απευθυντούμε στους φαρμακοποιούς. Η δουλειά της βιομηχανίας είναι να μην παρεμποδίζουμε την έρευνα. Το κείμενο πρέπει να βελτιωθεί διότι ε, πεκτεί κατά 10 με 12 χρόνια τον τρόπο με τον οποίο ε, μπορεί να παραταθεί η ζωή ενός φαρμάκου. Αυτό εμποδίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που παράγουν τα γενώσιμα να μπουν και αυτές στην αγορά. Δεν θέλουμε περιορισμένη πρόσβαση στα γενώσιμα. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ευζοίας των ζώων. Η κυρία Ντορνάνο. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, ε, των οποίων γύθηκε η Φρανσουάς Γκροστέτ και την οποία ευχαριστώ, Νομίζω ότι συζητούμε ένα κείμενο πολύ ευαίσθητο ακόμα. Παρόλους τους συμβασμούς πρέπει να εκφράσω τις δισταγμούς μου. Πρώτον, ε, ζώα τα οποία έχουν υποστεί κλινικές δοκιμές δεν θα πρέπει να καταναλώνονται. Ε, μια προφύλαξη σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Δεν πρέπει αυτός ο κίνδυνος ε, να περάσει στην τροφιμική αλυσίδα. Επίσης, η παραγωγή των κτηνιατρικών η υπόλοιψη των κτηνιατρικών φαρμάκων δεν πρέπει να γίνεται ε, στο ίντερνετ όταν αυτά πρέπει να συνταγογραφούνται και συνταγή θα πρέπει να χορηγούνται μόνο κτηνιάτρους ή κάτι αντίστοιχο. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τα δύο εξή. Ε, τον υγειονομικό κρίκο, τον οποίο εξασφαλίζουν οι κτηνιατροί, ε, και θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το επάγγελμα γιατί μέσω αυτών έχουμε μειώσει την κατανάλωση των, ε, των ε, αντιβιωτικών στη Γαλλία και δεύτερον δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε στην αύξηση της χρήσης πλαστών φαρμάκων εξαιτίας απορρίθμισης. Τέλος, ε, θα, δεν θα πρέπει να εξάγονται στην εσωτερική αγορά ζώα τα οποία τα φροντίζουν ε, επαγγελματίες που δεν είναι εκτινίατροι. Έχουμε δει σημαντικά προβλήματα με την απορρίθμιση των φαρμάκων. Ας είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί για το μέλλον. Σα Σας ευχαριστώ κύριο Σιλίζα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, δύο συγητές, κυρίως όμως την κυρία Φρανσουάς Γκοστέτ. Ε, να τη συγχαρώ γιατί πρόκειται για ένα πολύ τεχνικής φύσεως θέμα και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά ε, και μέσα στις διαπραγματεύσεις. Πολύ καλή έκθεση και πρέπει να την υπερψηφίσουμε όλοι μας. Ε, θα ήθελα να μιλήσω κυρίως ε, για την μικροβιακή αντοχή, την αντοχή στα αντιβιωτικά. Κάθε χρόνο πεθαίνουν 25.000 άνθρωποι επειδή τα αντιβιωτικά δεν είναι πλέον δραστικά και δεν βοηθούν τους ανθρώπους. Ε, και ε, αυτό ισχύει και για την κτηνιατρική. Ελέγχθησαν πάρα πολλά. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο όταν θα πάμε στον τριμερή διάλογο να δουν λιγάκι τις τροπολογίες 245 και 246 γιατί εκεί γίνεται λόγος όχι μόνο για το ότι θα πρέπει να καταγράψουμε τα αντιβιωτικά αλλά θα πρέπει να δούμε και τις συνέπειες ε, δηλαδή αυτό υπάρχει σε κάποια κράτη-μέλη και οι γεωργοί λένε ότι πριν έρθει ο γιατρός και μου πει τι πρέπει να κάνω ε, θα πρέπει να μου πείτε ε, πώς μπορώ να τα αποφύγω όλα αυτά δηλαδή τη χορήγηση ε, αντιβιωτικών με καλύτερη υγιεινή. Νομίζω αυτό πρέπει να ισχύσει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και κάτι άλλο για την ιατρική έναντι των ανθρώπων αν ε, πεθαίνουν ε, κάθε χρόνο τόσοι πολλοί άνθρωποι θα πρέπει να δούμε πού προσφέρεται η θεραπεία τους. Ε, η υγιεινή στα νοσοκομεία δεν είναι ικανοποιητική. Χρειαζόμαστε καινοτομίε. Ακόμα και αν είμαστε πολύ καλοί υπάρχουν, υπάρχει αυτό το θέμα της μικροβιακής αντοχής. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε την τροπολογία 22. Χρειαζόμαστε καινοτομία όχι μόνο στην κτηνιατρική αλλά κυρίως και στην ανθρώπινη ιατρική και παρακαλώ η Κομισιόν το συντομότερο δυνατόν να καταθέσει σχετική πρόταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπόρζαν για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τις σχέσεις ε, στη διανομή και τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων. Εγώ όμως θα εστιαστώ σε μία μονοπτυχή, την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιωτικά. Είναι σημαντικό που ο κανονισμό περιλαμβάνει διάταξη για την απαγόρευση συγκεκριμένων ε, αντιβιωτικών στα κτηνιατρικά φάρμακα, προκειμένου να τα κρατήσουμε μόνο για ανθρώπινη χρήση. Για να έχει όμω νόημα κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ισχύσει και αναδρομικά. Δηλαδή να συμπεριλάβει και την υποχρέωση απόσυρσης από την αγορά αυτών των αντιβιωτικών που θα κρατήσουμε για, τους, για ανθρώπινη χρήση και που ήδη κυκλοφορούν. Επίσης σημαντική είναι η σύνδεση της διανομής με τη συνταγογράφηση και μάλιστα από αρμόδιο άτομο. Επιπλέον όμως και για να αποτρέψουμε επιθενή ε, κακή χρήση ή κατάχρηση και για να εξυπηρετήσουμε, να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία θα πρέπει να απαγορεύσουμε τη διαδικτυακή πώληση αντιβιωτικών. Λόγω των διατροφικών συνηθιών μας και των εντατικών μεθόδων εκτροφής, η ανθρώπινη υγεία και η υγεία των ζώων είναι όλο και πιο λιλένδετες. Γι' αυτό το πρόβλημα των αντιβιωτικών θα πρέπει να το λύσουμε μέσω τη προσέγγιση μία και μοναδική υγεία. Ο κόδωνας του κινδύνου έχει χτυπήσει εδώ και πολύ καιρό, γι' αυτό και οι μελλοντικέ ε, ε, γενιές θα μας ρωτήσουν κάποια μέρα γιατί χάρη του κέρδους καταστρέψαμε ένα από τα σημαντικότερα ιατρικά επιτεύγματα στην ιστορία. Με αυτή την νομοθετική πρόταση έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να συμβάλλουμε στις παγκόσμιες προσπάθειες ε, για διαφύλαξη της αποτελεσματικότητας των αντιβιωτικών. Ε, επίσης ελπίζω ότι με τον κανονισμό αυτό θα συμβάλλουμε να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Σας ευχαριστώ κυρία Γκέρλινγκ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το μεγαλύτερο μέρος της ε, συζήτησης στο Κοινοβούλιο και τη συζήτηση ε, με το κοινό έχει περιστραφεί γύρω από τη μικροβιακή αντοχή. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό το θέμα και στενίζομαι την προσέγγιση της συγκήτριας σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της ε, προφυλακτικής χρήσης, τη προληπτικής χρήσης των αντιβιωτικών. Υπάρχουν όμως και άλλα σημεία στην έκθεση. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερος την εισηγητρία και του σκιώδη τους γιατί άκουσαν τις εκκλήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που ζήτησε να ε, διατηρήσει τις μακροχρόνιες ε, πρακτικές ε, για τη χρήση ή ατόμων με ειδικά προσόδια για την συνταγογράφηση. Φυσικά δεν λειτουργεί πάντα μία ενιαία λύση για όλους. Ιδιαίτερα στο υπόβαθρο της συζήτησης για το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι έχω και εγώ θετικά επιχειρήματα να προβάλλω. Επίσης, σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε για την απαγόρευση των μη ε, για το γενετικό στροποποιημένο οργανισμό θα οδηγούσε σε απόσυρση 19 ε, νέων ουσιών από τις ε, αγορές γιατί υπάρχει διάκριση μεταξύ των καλλιεργιών γενετικό τροποποιημένων ουσιών και των οργανισμών αυτών όταν περιέχονται σε φάρμακα. Ευχαριστώ Κύριο Χέιτεμα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται ότι μέσα σε μία γενιά η κατανάλωση των κανολικών θα, των αντιβιωτικών θα αυξηθεί κατά 67%. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη στις ε, προσπάθειές μας. Είναι ανεύθυνο να καλύπτουμε κάποια κενά στη θεραπευτική αγωγή με την εκτεταμένη χρήση αντιβιωτικών. Επίσης, η γενετική τροποποίηση θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται όπως ισχύει και για τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση. Γιατί χάρη στη γενετική τροποποίηση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να παραγάγουμε την ισουλίνη που είναι απαραίτητη για το διαβήτη. Και μάλιστα μερικές φορές η Σουλήνη είναι η μόνη δυνατότητα που έχουν οι διαβητικοί. Όσοι θέλουν να απαγορεύσουν τη γενετική τροποποίηση ε, στα φάρμακα διακυβεύουν την υγεία και των ζώων και των ανθρώπων και δεν έχουν και κανένα έρισμα για να στηρίξουν τα επιχειρηματά τους. Ο κανονισμός ε, αυτός έχει θετικές ε, πτυχές εξασφάλιση ασφαλών και προσβάσιμων κτηνιατικών φαρμάκων για όλους. Ε, το θέμα της μικροβιακής αντίστασης, το ΙΤΟ και των μικρών αγορών επίσης είναι πτυχές οι οποίες ρυθμίζουν σωστά. Θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα πιο μακριά αν δεν είχαν πιέσει οι πολυεθνικές εταιρείες που θέλουν να διατηρήσουν τα προνόμια τους και να ε, ε, αυξήσουν τα κέρδη τους. Ε, για τις μικρές ε, χώρες ε, θα ήταν πιο χρήσιμο να γίνει πιο κεντρική η αδειοδότηση. Η καλή εφαρμογή δεν λύνεται, η καλή χρήση δεν λύνεται μόνο με αυτόν τον κανονισμό. Χρειάζεται μια κοινή αγροτική πολιτική διαφορετική που αυτή τη στιγμή προάγει την μονοκαλλιέργεια. Ευχαριστώ. Thank you. Madam Scott Κυρία Σκοτ Κάτω. Ένα λεπτό. Ο σύνδεσμος ανάμεσα στη χρήση των ε, αντιβιωτικών και την αύξηση της μικροβιακής αντοχής είχε καταδειχθεί. Ε, ο, ε, ο Βρετανός επιστήμονας είπε ότι η, η μεγαλύτερη χρήση των αντιβιωτικών στα ζώα θα αυξήσει τη θνησιμότητα στους ανθρώπους αργότερα. Ε, η αύξηση της μικροβικής αντοχής είναι δεδομένη και γι' αυτό λόγο πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών και στους ανθρώπους και στα ζώα. Αυτή τη στιγμή τα αντιβιωτικά μπορούν να, συνταγοραφηθούν να συνταγογραφηθούν σε όλα τα ζώα, ακόμα και αν δεν νοσούν, ε, μόνο επειδή έχουν κάποιο κίνδυνο να μολυνθούν. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη χρήση των αντιβιωτικών. Ως ε, πράσινοι Πιστεύουμε ότι η χρήση των αντιβιωτικών δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις καλές πρακτικές. Όταν τα ζώα βέβαια διατηρούνται ε, σε μεγάλες πυκνότητες, σε συνθήκες υγιεινής που δεν είναι καλές, είναι προφανές ότι αυξάνεται ο κίνδυνος και χρειάζονται αντιβιωτικά. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις συνθήκες και όχι να αυξήσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρίδη για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, στο, το UKIP πιστεύει ότι η, χρήσιμη, η, η υπεύθυνη χρήση των αντιβιωτικών είναι πολύ σημαντική στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδιαίτερα αυτά που χρησιμοποιούνται στα ζώα μα. Είναι πολύ σημαντικό όμω η, είναι πολύ οι γεωργοί να διατηρούν την υγεία των ε, ζώων ε, και την ποιότητα των προϊόντων για την οποία είμαστε γνωστοί. Όμω τα κτηνιατρικά φάρμακα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την, ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της, ε, ε, της ποιότητας ε, ή ναι, την υποκατάσταση των καλών συνθήκων εκτροφής. Η νομοθεσία αυτή τη στιγμή που ισχύει από το 2001-2004 στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδιαίτερα αύξηση του κόστους εξαιτία του διοικητικού άχθους που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες. Γι' αυτό το λόγο διαφωνούμε με την δημιουργία ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου Πιστεύουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Μόνο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έπρεπε να έχει την αρμοδιότητα να νομοθετήσει αυτό το θέμα και όταν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα το κάνει. Ευχαριστώ. Κυρία Γκαρντίνη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους δύο συγητές, την κυρία Γκροστέτ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά ε, Ευχαριστώ βεβαίω και όλου του άλλου και του συναντέλφου ε, που παρένεψαν. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Αύριο θα ψηφίσουμε και κατ' ουσίαν θα κάνουμε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση τροποποίησης της διαδικασίας με την οποία αντιοδοτούν τα φάρμακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, ψηφίζοντας τις ε, τροπολογίες του κανονισμού μπορούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα προς την ε, ριζική ε, μείωση, εύχομαι, του χρόνου που περνά από τη στιγμή που εγκρίνεται ένα νέο φάρμακο μέχρι ε, να φτάσει να ε, τεθεί σε ισχύ, να αρχίσει να Ε, Αυτό που ενδιαφέρει είναι ο χρονισμός. Το ίδιο φάρμακο πολλές φορές ε, αξιολογείται για το κατά πόσο είναι δραστικό 28 φορές σε 28 διαφορετικά κράτη-μέλη. Κλασική είναι η περίπτωση που είναι γνωστή η περίπτωση του τρανσουδίου Zumap ενό ειδικού φαρμάκου ε, για τον καρκίνο του στήθους και ήταν ιδιαίτερα δραστικό κρίθηκε, συμπεριλήφθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όμως για να φτάσει το φάρμακο αυτό σε ορισμένα κράτη-μέλη για να αρχίσει να πωλείται. πέρασαν μέχρι και 10 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει πια να ανοίξει ένας καινούριος δρόμος για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες. Κυρία Μελιόρα, ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε εδώ ένα πολύ σημαντικό κανονισμό και υπόθηκα πάρα πολλά για ένα θέμα που με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ, για τα αντιβιωτικά. Εγώ όμω όλα αυτά όσα θα τα επαναλάβω και θα πω με απόλυτη σαφήνεια. Κοιτάξτε, τα αντιβιωτικά δεν είναι παχυντικό ούτε είναι υποκατάστατο κτίνο ε, κτηνοτροφίας Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε κατά νου. Τα εφεδρικά αντιβιωτικά νομίζω ήδη από την ονομασία καθίσατε σαφές ότι τα εφεδρικά θα πρέπει να φορούν τον άνθρωπο. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ για το ότι στον κανονισμό προβλέπεται αυστηρός έλεγχος ε, για όλα τα κράτη-μέλη θα αναφέρετε ότι πρέπει να καταγράφεται η χρήση των αντιβιωτικών και χαίρομαι επίσης πάρα πολύ και ευχαριστώ τους εισηγητές ε, για το ότι έχουν ε, αξιολογηθεί και επιπτώσει στο περιβάλλον από την παραγωγή μέχρι το να εντοπίσουμε υπολείμματα στο χωράφι τώρα πια μπορούμε να γνωρίζουμε ποιε είναι οι επιπτώσεις του περιβάλλον και τι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ όλους σας. Νομίζω κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος για να ε, αντιμετωπίζουμε τα την ιατρικά φάρμακα με διαφορετικό τρόπο. Ο κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως και ο των μεταρρυθμιστών συντηρητικών από την Επιτροπή Γεωργίας θεωρώ αυτή την έκθεση για τα κτηνιατρικά φάρμακα πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την έρευνα για νέα κτηνιατρικά φάρμακα. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε και οι περίοδοι εφαρμογής να είναι σωστές και φυσικά να ελαφρύνουμε με αποτελεσματικό τρόπο το γραφειοκρατικό άκτο για να μπορέσουν οι εταιρείε να, κάνουν, να, να ζητάνε αποκεντρωμένα τις άδειε θέσεις εμπορία και να λειτουργούν αποτελεσματικά. Η προφυλακτική χρήση των αντιβιωτικών δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από κοινού. Είναι σημαντικό να έχουμε κοινή προσέγγιση και χαίρομαι που το κείμενο το επισημαίνει. Σε μερικές χώρες περιορίστηκε η χρήση των αντιβιωτικών, κάτι που είναι ευπρόσδεκτο, αλλά αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί σε κοινοτικό στόχο. Θα πρέπει όλοι να κάνουμε προσπάθειες και να περιορίσουμε τα αντιβιωτικά πανευρωπαϊκά για να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική που θα αποφέρει καρπούς. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριο Φέντερλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το βήμα που πραγματοποιούμε σήμερα είναι πολύ σημαντικό σε ένα μακροχρόνιο αγώνα μας. Ο κύριος Όρσεν και μία άλλη συνάδελφος από τους φιλελεύθερους Σουηδου ξεκίνησε τον αγώνα αυτό τη δεκαετία του 90. Τότε ήδη μιλούσαμε για ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και διαπιστώνουμε ότι όλα τα κόμματα χαιρετίζουν την πρόταση, κάτι που σημαίνει ότι όντως παραδέχονται την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και θα φανεί ε, και αργότερα στη συζήτηση για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Είναι πολύ σημαντικό πώς αντιμετωπίζουμε την υγεία. Φυσικά τα αντιβιωτικά θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά. Γι' αυτό θα πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση τους. Φυσικά, χάρη στα αντιβιωτικά η πνευμονία δεν είναι πια θανατηφόρα ασθένεια. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να φροντίσουμε να καταπολεμήσουμε τη μικροβιακή αντοχή για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη υγεία των ζώων και των ανθρώπων και να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίνς για 1,5 λεπτό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 Κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτριά μας, την κυρία Γκροστέτ, ε, γιατί πραγματικά κατέθεσε μια θαυμάσια έκθεση. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα δραστικά φάρμακα για τα ζώα, το να υπάρχουν αυτά τα φάρμακα ε, και να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή, αυτός είναι ο στόχος αυτού του πακέτου. Είμαι σίγουρος ότι ε, μπορούμε πολλά να καταφέρουμε ε, θα υπάρχει καλύτερη έρευνα και θα ε, περιοριστεί η χρήση των αντιβιωτικών. Και η προληπτική χρήση αντιβιωτικών θα περιοριστεί στο ελάχιστο. Ε, θα απαγορεύεται πλήρως να χρησιμοποιούνται τα αντιβιωτικά ως μια καθημερινή ρουτίνα για τα οικόσιτα ζώα μας, για να έχουμε σωστή θεραπεία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλου είδους πρακτικές, την ομοιοπαθητική, γιατί όχι. Τα υποθετικά φάρμακα παίζουν σημαντικό ρόλο. Εγώ διαφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως από την ομάδα ECR. Τέλος, όσον αφορά τον περιορισμό ε, της ε, μικροβιακής αντίστασης, ε, η αντοχής, τα μειοπαθητικά μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Για μένα λοιπόν πρέπει ο κανονισμός αυτός να συνδυαστεί με τον κανονισμό για τις ζωοτροφές και αυτά να αντιμετωπίζονται ως ένα πακέτο. Γι' αυτό λοιπόν Χαίρομαι που κατέστη δυνατό να καταθέσουμε αυτή την πρόταση γιατί ενισχύουμε το ρόλο του κτηνέατρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκούτελαντ, ένα Η αυξημένη μικροβιακή αντοχή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε μελετήσει επαρκώ ω τώρα. Οπότε η έκθεση αυτή είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μολύνσει οι οποίε έχουν, που προκαλούνται από ανθεκτικά μικρόβια γίνονται όλο και πιο δύσκολο να θεραπευτούν και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Ε, βλέπουμε τι συνέπειε του καθημερινά στα παιδιά και στα βρέφη, ε, στους ηλικιωμένους, σε νεογνά κλπ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν χρειαζόμαστε ένα, μια ισχυρή νομοθεσία για να ενισχύσουμε την ε, καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς, δεν θέλουμε την τακτική και περιττή χρήση, προφυλακτική χρήση ε, αντιβιωτικών στα ζώα. Τα αντιβιωτικά θα πρέπει να δίδονται σε ζώα που νοσούν μόνον. Και με αυτή την ε, νομοθεσία νομίζω παίρνουμε, κάνουμε ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Τελικά όμως θα πρέπει να απαγορεύσουμε την προφυλακτική χρήση των αντιβιωτικών στα ζώα. Ευχαριστώ. Κυρία Γιούσο για ένα μισή λεπτό. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την συνάδελφο κυρία Γκροστέτ ήταν τεράστιος ο αριθμός των προτάσεων τροπολογίας ε, με, ε, με το ε, πνεύμα συνεργασία που έδειξε τα καταφέραμε. Έπρεπε να κάνουμε διάκριση ε, ανάμεσα στους διάφορους τύπους αγωγής προφυλακτικό, θεραπευτικό και μεταφυλακτικό. Θα πρέπει να μειώσουμε επίσης το διοικητικό άχθος και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε επαρκείς ε, εγγυήσεις για την ασφάλεια ε, και την, την ενημέρωση σε ό,τι φορά τη χρήση. Για την ε, διαθεσιμότητα δεν είναι ίσον σημασία ζήτημα. Πρέπει να βρούμε λύση για συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένε νόσους τι οποίε ονομάζουμε ίσονο σημασία χρήση και νόσου. Ε, θα πρέπει επίσης να στηρίξουμε τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της καινοτομίας. Τέλος, τροποποιήθηκε η πρόταση ό,τι αφορά την δυνατότητα κτηνίατροι να χρησιμοποιούν ε, φάρμακα για ενδείξεις και είδη που δεν προβλέπονται από τις ε, συστάσεις του κατασκευαστή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα σύστημα συνταγογράφησης ε, χιονοστιβάδας ε, και να χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό θα πρέπει βέβαια να το κάνει ο κτηνίατρος. Ευχαριστώ. Thank you. Madame um, one minute. Κυρία για ένα λεπτό. κυρία Σαλντεμόζε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ αξιόλογη έκθεσή της, ε, την οποία και ε, θα υπερψηφίσω ολόθερμα. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε σοβαρά με το θέμα της μικροβιοικής αντοχής στα αντιβιωτικά σε μια κοινοτική νομοθεσία. Και είναι σημαντικό γιατί 25.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας της μικροβιακής αντοχής. Επειδή τα αντιβιωτικά δεν είναι αποτελεσματικά για τις λοιμώξεις τους. Και αυτό οφείλεται στην υπερβολική χρήση των αντιβιωτικών στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση ο κανονισμός αυτός. Πλησιάζουμε στην ολοσχερή ε, απαγόρευση της προφυλακτικής χρήσης των αντιβιωτικών. Δεν μπορούμε να συνταγογραφούμε αντιβιωτικά για υγιή ζώα. Μόνο ζώα που είναι άρρωστα θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή. Και φυσικά η συνταγογράφηση να γίνεται από τους αρμοδίους Ελπίζω την επόμενη φορά είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι, πάντως πάλι καλά που έστω και καθυστερημένα ασχολούμαστε με τη μικροβιακή αντοχή. Ο κύριος Βαντεγκέντελαρ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτρόπε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω του ηγητέ μα για τι εξαιρετικέ του εκθέσει. Επιτέλους, ε, προσπαθούμε να βρούμε ένα αποτελεσματικό τρόπο για να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για νομοθετικές διατάξεις που θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε τη μικροβιακή αντοχή. Ένα ιδιαίτερα προβληματικό ζήτημα. Θα πρέπει να καινοτομήσουμε και να επενδύσουμε σε έρευνα σε νέα φάρμακα και να μειώσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών. Φυσικά δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε όλο χερό τη χρήση τους. Αυτό θα ήταν υπερβολικό, αλλά σίγουρα να την περιορίσουμε Θέλουμε υπεύθυνη και προσεκτική χρήση αντιβιωτικών φαρμάκων και νομίζω ότι η έκθεση υιοθετεί τη σωστή προσέγγιση και προτείνει μια μερική απαγόρευση των πωλήσεων μέσω διαδικτύου, για παράδειγμα, ή την προφυλακτική, απαγόρευση της προφυλακτικής χρήσης. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε την περαιτέρω επέκταση της μικροβιακής αντοχής. Θα πρέπει να συσπηρωθούμε, να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες, να επιτρέψουμε τη διατήρηση της χρήσης των αντιβιωτικών, αλλά μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Φυσικά ε, θα πρέπει να έχουμε και ένα κατάλογο εξαιρέσεων, αλλά αυτό θα το καταρτήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα στηρίζεται σε επιστημονικά πορίσματα. Η κυρία Γιλέρα Γαρσία έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω τη φωνή μου στα συγχαρητήρια στους δύο εισηγητές, την κυρία Γκροστέτ φυσικά για το τιτάνιο έργο που επιτέλεσε, αλλά και στον κύριο Τανασέσκου. Νομίζω ότι γενικώ ε, επιτελέσαμε ένα πολύ αξιόλογο έργο, δεδομένης της δυσκολίας και του τεχνικού χαρακτήρα του κανονισμού. Εγώ είμαι η για τις φαρμακούχες ζωοτροφές αρμόδια κατ' ουσία για την έκθεση αυτή είναι η Επιτροπή Γεωργίας. Ακριβώς ε, ε, λόγω της συνάφειας αυτής της έκθεσης με την έκθεση τη κυρίας Γκροστές παρακολούθησε εκ του σύνεγγες και τη δική της έκθεση και θα ήθελα να την ευχαριστήσω θερμά για το έργο της γιατί μας διευκόλυνε ε, και στη δική μας έκθεση για τον κανονισμό για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Ένας κανονισμός που θα ρυθμίσει τον τρόπο χορήγησης των κτηνιατρικών φαρμάκων είναι πολύ σημαντικό. Και στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ε, την ψηφοφορία στην Επιτροπή Γεωργίας και της δικής μου έκθεσης για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Έχουμε δυσκολίες για να βρούμε κτηνιατρικά φάρμακα για τα είδη ίσονα σημασία όπως τα προκαλούμε Και χαίρομαι που ε, υιοθετήσαμε αυτή τη διαδικασία αν κασκάτ όπως πρότεινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος που βελτιώνει κατά πολύ την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην διαδικασία Catch the Eye. Καπισόν ε, Λουίς. Ευχαριστώ. Η μικροβιακή αντίσταση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσια υγεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο. Ας λάβουμε όλα τα μέτρα που διαθέτουμε. Γι' αυτό το λόγο θέλω να συγχαρώ τους συγγητές γιατί κατάφεραν και έκαναν το κείμενο της Κομισιόν πιο φιλόδοξο. Εποφελήθηκαν λοιπόν της ευκαιρίας. Έχει βελτιωθεί προφανώς το κείμενο πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό βήμα ε, προκειμένου να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της μικροευαϊκής αντοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 25.000 νεκροί το χρόνο και πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά που προέρχεται από τη μικροβιακή αντοχή. Υπάρχει βέβαια πράγματα που μπορούν να γίνουν στο μέλλον και είμαι σίγουρη ότι θα, το θα τα κάνουμε. Όμως ε, η πορεία ξεκίνησε. Συγχαίρω λοιπόν και εγώ τους συνεισηγητές και ελπίζω ότι αυτό αποτελεί απλώς την εκκίνηση. Ε, κυρία Τιβαζή, συγχαρητήρια στην κυρία Γκροστέτ ε, Πολύ σημαντικό το έργο της, ήταν ε, πολύ δεκτική. Πρέπει ασφαλώς να μειώσουμε την ε, μικροβιακή αντίσταση, διότι η χρήση των αντιβιωτικών συνδέεται με την αύξηση της μικροβιακής ε, αντίστασης. Ε, ο περιορισμός της ε, πώληση των αντιβιωτικών μέσω του ίντερνετ ε, κλπ. Η, η, η, χρήση των αντιβιωτικών μόνο γενικά, ναι, η χρήση των αντιβιωτικών μόνο για μεταφυλακτική δράση και η διατήρηση ορισμένων ειδών για ανθρώπινη χρήση είναι πολύ σημαντικά μέτρα. Πρέπει όμως να έχουμε και αναλλακτικές λύσεις. Μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών. Όμως, θα πρέπει ταυτόχρονα να ενισχύσουμε και εδώ στηρίζω την ε, τροπολογία Όσλινγκ την ομοιοπαθητική. Και επίσης θα πρέπει να αυξήσουμε ε, την έρευνα ε, για τα για τους βακτηριοφάγους που μπορούν να καταπολεμήσουν ορισμένες ασθένειες. Επίσης θα πρέπει να δούμε τη χρήση των αντιβιωτικών στη θάλασσα, όπως για παράδειγμα στην εκτροφή Σολομού. Εκεί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθόλου. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τα κτηνιατρικά φάρμακα απαιτεί να υπάρχουν βελτιώσει όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Έχουμε το φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής, λείπουν κίνητρα για καινοτομία και υπερβολική γραφειοκρατία στην φαρμακοεπαγρύπνηση. Ε, πολλά κενά πρέπει να καλυφθούν. Το βασικό πρόβλημα αναμφίβολα είναι η μικροβιακή αντοχή. Έτσι λοιπόν απολύτως απαραίτητο τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τους ε, τις οδηγίες ε, για τη χρήση των αντιβιωτικών. Ε, υπάρχουν πολλά περίπλοκα στοιχεία για τη χρήση αντιβιωτικών, είναι όμως απαραίτητα για να υπάρχει σωστή χορήγηση για λόγους προφύλαξης. Η μικροβιακή αντοχή βλέπουμε ότι είναι κυρίως συνδεδεμένη με την ανθρώπινη χορήγηση. Θα πρέπει να είναι λοιπόν πιο περιορισμένη η δυνατότητα χορήγησης ε, για τους κτηνιάτρους να χορηγούν φάρμακα. Η λύση είναι να επανέλθει η αρχή όπου όταν διαφυλάσσουμε την υγεία του ζώου διαφυλάσσουμε και την υγεία του ανθρώπου. κύριος Μαριάς παρακαλώ πρόεδρε συζητούμε για τη χορήγηση αδείας για τα φάρμακα που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση καθώς και για τις επιπτώσεις των φαρμάκων αυτών στη δημόσια υγεία. αρχικά όσον αφορά την κεντρική άδεια κυκλοφορία για κτηνιατρικά προϊόντα θα πρέπει να αποσυνδεθεί από εκείνη των φαρμάκων για τους ανθρώπους καθώς οι ανάγκες του κτηνιατρικού τομέα για φάρμακα διαφέρουν κατά πολύ από τις ανθρώπινες. άλλωστε στον κτηνιατρικό τομέα υπάρχουν διαφορετικά είδη ζώων με αποτέλεσμα να δημιουργείται κατακαιρματισμός της αγοράς και να αυξάνεται η ανάγκη για επενδύσεις προκειμένου να επεκταθεί η έγκριση φαρμάκων από το ένα είδος ζώο στο άλλο. επιπλέον παρά τα υγειονομικά μέτρα που λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι τα ζώα χρειάζονται και κτηνιατρικά φάρμακα για να αντιμετωπίσουν μια νόσο και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη μετάδοσή της στον άνθρωπο. επομένως η κτηνιατρική βιομηχανία οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι φαρμακευτικές ουσίες που διατίθενται στην αγορά δεν είναι επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία για την υγεία των ζώων και των περιβάλλων και θα πρέπει επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα αντιβιωτικά που χορηγεί σε ζώα που προορίζονται για παραγωγή τροφίμων. ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Μπούχνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Ε, πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για το ότι έρχεται ένας ε, κανονισμός ε, ο οποίος κάνει κάτι για την μικροβιακή αντοχή. Να σας υπενθυμίσω ότι στη Γερμανία περίπου το 88% της, του κρέατος γαλοπούλας που πωλείται στα σούπερ μάρκετ επιβαρύνεται με μικροβιακή αντοχή. Πώς μπορούμε όμως ε, να τα απαγορεύσουμε όλα αυτά όπου έχουμε κτηνοτροφικές μονάδες με εκατοντάδες χιλιάδες ε, πουλερικά. Για τέτοιου είδους λοιπόν πουλερικά χρειαζόμαστε τα αντιβιωτικά. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ θερμά αύριο ε, που θα εγκρίνουμε αυτό τον κανονισμό που είναι πάρα πολύ καλός να μην εφησυχάσουμε αλλά να έχουμε κατά νου ότι ο αγώνας θα είναι σκληρός να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός και να τον υπερασπιστούμε από επιθέσεις εκ των έξω. Κλείνει λοιπόν η διαδικασία Catch the Eye ε, και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κ. Αντρουκάητης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ακούσατε τις εξηγήσεις που έδωσα ε, παρουσιάζοντας τις ε, προτάσεις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για αυτή τη νέα πρόταση σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα και άκουσα εγώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις σας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε συμφωνία σε αυτούς τους νέους κανόνες για να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα κτηνιατρικών φαρμάκων και αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που από τη χορήγηση αντιβιωτικών κατά την εκτροφή των ζώων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να υπάρχουν και άλλες διατάξεις. Οι περισσότερες εξ αυτών που συζητήθηκαν είναι θετικές. Επίσης ε, χαιρετίζω την τροπολογία που αναφέρει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την προφυλακτική χρήση και την μεταφυλακτική χρήση των αντιβιωτικών. Η πρώτη αφορά μεμονωμένα ζώα ε, και δικαιολογεί απόλυτα από τον κτηνίατρο. Η δεύτερη αφορά ε, ζώα που είναι σε κλινική θεραπεία και μεμονωμένα ζώα που ε, θεωρούνται ότι είναι υψηλός φορέας ε, κινδύνου για μετάδοση της νόσου. Νομίζω έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου και κατέστη δυνατόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Βεβαίως υπολείπονται ακόμα αρκετά σε σχέση με την καινοτομία και τη χρήση νέων καινοτόμων θεραπείων. Αυτό επιτρέψτε μου να πω είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Καινοτομία λοιπόν, πρόσβαση σε εκτινιατρικά φάρμακα, αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, προστασία της δημόσιας υγείας, αυτά δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους. Κάθε άλλο η καινοτομία είναι το βασικό εργαλείο για να μπορούμε να εγγυητούμε την δημόσια υγεία. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι ε, πρέπει να συζητήσουμε σε βάθος και κάποια άλλα θέματα όπως την πρόταση να συγκεντρώνονται δεδομένα και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Αυτό πρέπει να εξηγηθεί περαιτέρω γιατί είναι δυνατόν να ε, συνεπάγεται διοικητική επιβάρυνση. Είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι λόγω της πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε στο εγγύς μέλλον να επιτύχουμε το στόχο μας. Για άλλη μια φορά κυρία Γκροστέτ και κύριε Τόμασέ Λουτσέσκου Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά σας. Και τώρα πλέον έχει έρθει η στιγμή του ε, Συμβουλίου να ακολουθεί το Συμβούλιο το καλό παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιταχύνει τις εργασίες του έτσι ώστε να φτάσουμε στην πρώτη ανάγνωση. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω για την ανεπιφύλακτη υποστήριξη της Κομισιόν θέλουμε να επιτευχθεί ε, το συντομότερο συμφωνία με το Συμβούλιο. Ωραία, επιστρέφω στους εισηγητέ. Κύριε Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που παρνέβησαν στη συζήτηση σήμερα το βράδυ. Να του ευχαριστήσω για τη στήριξή τους. Εν γέννη και εν συνόλο ε, βλέπω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο της έκθεσης. Όμω, αυτό το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα συλλογική εργασία. Δεν είναι μόνο η δική μου η έκθεση, είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό το λόγο θέλω να συγχαρώ όλου και όλου οι ηγητέ, ιδιαίτερω αυτούς που γιατί συμμετείχαν σε πολλές συναντήσει το αντικείμενο ήταν πολύ περίπλοκο συχνά. Έπρεπε να λάβουμε υπόψη τι ιδιαιτερότητε κάποιων χωρών, λαμβάνοντα υπόψη τι κατευθείαν γραμμέ που ήταν στην πραγματικότητα, όπω είπαμε, καταπολέμηση τη μικροβιακή αντοχής. Δεν θα επανέλθω στι λεπτομέρειε. μίλησε ο επίτροπο, είναι πολύ σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα θέλαμε να στηρίξουμε και την καινοτομία. Γιατί εκεί ε, έχουμε έλλειψη εκτινετρικών φαρμάκων ε, Γι' αυτό το λόγο προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής και την ε, καινοτομία, την πρόθεση καινοτομίας. Θέλουμε ε, εμπορικά προϊόντα διαφορετικά για ίσονος ή μίζωνος σημασίας ε, ζώα, ακόμα και για ιδιαίτερα όντα ζώα όπως οι μέλισσες. Για τις μέλισσες έχουμε ειδικά προβλήματα. Για αυτό το λόγο ζητούμε προστασία 20 ετών. Για την ε, πώληση μέσω διαδικτύου επιτρέπεται, αλλά όχι για τα αντιβιωτικά, όχι για τις ψυχότροπες ε, ουσίες. Ε, προσπαθούμε να δούμε, προσπαθήσαμε να δούμε τι είναι το σημαντικό και αυτό να προωθήσουμε. λάβουμε υπόψη επίσης το περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Το είπαν οι συνάδελφοί μας. Αν έχω ένα μήνυμα να στείλω, είναι ε, ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή πλειοψηφία στην ψηφοφορία. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πιέσουμε το Συμβούλιο. Να μην χάσουμε ούτε ένα λεπτό και να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ο φόβος που έχω είναι ότι το Συμβούλιο ε, θα βάλει λίγο στο περιθώριο το θέμα αυτό, θα το αμελήσει και ότι θα καθυστερήσουμε. Κάτι τέτοιο ε, είναι, θα ήταν σοβαρό πρόβλημα γιατί πρόκειται για ένα θέμα υγείας των ζώων, υγείας, ε, ανθρώπινης υγείας. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν στηρίξτε μαζικά την πρόταση αυτή έτσι ώστε να πιέσουμε το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τανασέσκου, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα την κυρία Γκροστέτ και τους ε, σκιώδεις εισηγητές ε, για την δουλειά που έχουν κάνει εδώ πέρα και την εξαιρετική συνεργασία. Να τονίσω το ότι με τις ε, εκθέσεις αυτές έχουμε πλέον ξεκάθαρη νομοθεσία που ταιριάζει καλύτερα στον κτηνιατρικό τομέα. Ξεκαθάρισε και ο ρόλος της υπηρεσίας στην αδειοδότηση των φαρμάκων και η αυριανή ψηφοφορία είναι ένα μεγάλο βήμα για να προστατεύσουμε την υγεία ανθρώπων και ζώων και βεβαίω για να καταποντιμήσουμε την ε, αντοχή στα αντιβιωτικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Κλείνει εδώ η κοινή συζήτηση. Το θέμα θα το ψηφίσουμε αύριο.